Δεν προβλέπεται η διαδικασία catch the eye, ούτε θα γίνουν δεκτές ερωτήσεις με ε, γαλάζια κάρτα. Έχει το λόγο εξ ονόματος του Συμβουλίου η κυρία Τζάντα Ζανίνα Λουκατσέβικ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Πριν περάσω στην ημερήσια διάταξη αυτή καθεαυτή πρέπει να σας πω ότι είναι η τελευταία ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό Λετωνική Προεδρία. Και είναι η μέρα που η χώρα μου γιορτάζει το αποκορύφωμα του καλοκαιριού. Προκειμένου λοιπόν να τιμήσουμε την ημέρα αυτή και μια που έχουμε και την τελική αυτή προεδρία θα μιλήσω στα λετωνικά. Ολοκληρώνεται λοιπόν η Λετωνική Προεδρία σήμερα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με αυτή την τελευταία ολομέλειά του. Η ημερήσια διάταξη στην σύνοδο του Συμβουλίου είναι πυκνή. Οι επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων θα αποφασίσουν για τη μετανάστευση, για την ασφάλεια, και για την οικονομική διακυβέρνηση. Πριν λοιπόν περάσουμε σε λεπτομέρειες, θέλω να σας ενημερώσω για την άτυπη συνάντηση στην Ευρωζώνη επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων μετά από πρωτοβουλία του Πρόεδρου Τάσκ. Στόχος ήταν να έχουμε περισσότερη σαφήνεια όσον αφορά την κατάσταση στην Ελλάδα. Οι επικεφαλείς κρατών και κυβερνήσεων αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα και συζήτησαν και την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και τους διεθνείς πιστωτές. Στη συνάντηση αυτή ο κύριος Τάσκε θέλει να αλλάξει τη δυναμική των διαπραγματεύσεων και να της δώσει μια νέα θετική όθηση. Η συνάντηση της Δευτέρας πράγματι έδωσε αυτή τη θετική όθηση. Όπως είπε και ο ίδιος ο πρόεδρος Τάσκα, σε συνδυασμό με τους διεθνείς πιστωτές υπάρχει μια νέα προσέγγιση της ελληνικής κυβέρνησης που πάει προς τη σωτή κατεύθυνση. Τώρα πρέπει να ακολουθήσει η δράση. Ο Πρωθυπουργό Τσίπρας και οι διεθνείς πιστωτές δουλεύουν από κοινού μαζί ώστε σήμερα το βράδυ στη συνάντηση του Eurogroup να έχουμε αποτελέσματα μετά από τη δουλειά που έχει γίνει όσον αφορά το μεταρρυθμιστικό σχέδιο που θα υποβληθεί έτσι αύριο στους επικεφαλείς κρατών και κυβερνήσεων. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, για να επανέλθουμε τώρα στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Επιτρέψτε μου να αρχίσω με τη μετανάστευση. Θα είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που θα συζητηθούν αύριο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά, ήδη τον Απρίλιο του 2015 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε απόφαση για έκτακτα μέτρα προκειμένου να αποφύγουμε επιπλέον θανάτου στη θάλασσα και προκειμένου να βρούμε νέους τρόπους να αντιμετωπίσουμε ε, το θέμα αυτό της παράνομης διακίνησης ανθρώπων. Και το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπε ότι τα αποτελέσματα εκείνα του Συμβουλίου δεν ήταν επαρκή. Ήδη λοιπόν τώρα θέλω να σας πω ότι στόχος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τότε δεν ήταν να λύσει όλα τα δυνάμει προβλήματα της μετανάστευσης. Συνεπώς δεν υπάρχουν γρήγορες και βιαστικές λύσεις. Μακροπρόθεσμες λύσεις μπορούν να βρεθούν μόνο εφόσον έχουμε μια στοχευμένη και συνολική προσέγγιση που θα εφαρμόζεται σταδιακά. Αύριο η συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα είναι ακριβώ το επόμενο βήμα προκειμένου να εφαρμόσουμε την προσέγγιση αυτή. Στου λίγου μήνες που πέρασαν από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν συνεισφέρει προς την εξέβρεση λύσης. Και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και το Συμβούλιο έδωσαν ένα χάρτη πορείας στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να προχωρήσει βάση αυτού. Και υπάρχει και έκθεση όσον αφορά τη μετανάστευση. Ήδη το Συμβούλιο λοιπόν άρχισε να δουλεύει πάνω στις διάφορες αυτές πτυχές και προσπαθεί να εφαρμόσει τα όσα αναφέρονται στο πρόγραμμα για τη μετανάστευση. Αύριο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα σημειώσει τρία πράγματα. Πρώτον, το θέμα της επαναγκατάστασης. Το θέμα της επιστροφής, της επανεισδοχής δηλαδή. Και τρίτον, το θέμα της συνεργασίας με τις χώρες προέλευσης και τις χώρες transit. Όλα αυτά βέβαια είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και μια συνολική προσέγγιση μας επιτρέπει να προστατεύσουμε αυτούς που περισσότερο χρειάζονται την προστασία μας. Βέβαια επαναλαμβάνω, δεν φτάνουν αυτά συγχρόνως πρέπει να έχουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα επιστροφής των ε, μεταναστών. Δεν είναι εξάλλου κανένα μυστικό. Συνεχίζονται οι συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την μετακατάσταση των ε, προσφύγων. Χτες οι συζητήσεις που είχαμε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων έδειξαν ότι χρειάζεται συνένεση προκειμένου να επιτευχθεί λύση για το μεταναστευτικό. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στην αλληλεγγύη και την υπευθυνότητα. Είναι κομμάτια της μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Υπουργοί έδειξαν ότι είναι έτοιμοι να δείξουν την αλληλεγγύη τους, να βρουν λύση προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό. Αναφίβολα χρειάζεται ο κατάλληλος μηχανισμός ο οποίος θα μας επιτρέψει να δώσουμε μια απάντηση σε αυτήν την έκτακτη κατάσταση και που θα βοηθήσει συγχρόνως τις χώρες εκείνες που πρώτες από οποιαδήποτε άλλη αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις των μεταναστευτικών αυτών ορών. Πολιτικά και τεχνικά τα ζητήματα. Οι απόψει των χωρών μελών βέβαια διαφέρουν για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιο θα πρέπει να είναι ο ρόλο των χωρών μελών. Συνεπώ, πρέπει να κάνει περισσότερα ακόμα το Συμβούλιο πριν ληφθούν νέε αποφάσει. Πάντω, η μετανάστευση είναι ευαίσθητο ζήτημα. Απαιτεί ισορροπημένη προσέγγιση. Δεν μπορεί έτσι στα γρήγορα να βρεθεί κάποια λύση. Η Ουγγαρία, μάλιστα, μάθαμε ότι μονομερός σταματά την εφαρμογή του συστήματος Δουβλίνο 2. Μονομερείς δράσεις δεν είναι λύση. Μόνο με διάλογο και με αποκοινού δράση μπορούμε να εφαρμόσουμε καλά το κεκτημένο και να βρούμε λύσεις στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Χρειάζεται συνολική προσέγγιση. Αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί μόνο τότε μπορούμε να έχουμε συνολική στήριξη. Και έτσι να καταλήξουμε σε λύσεις μακροπρόθεσμα. Πάντως, οι προκλήσεις της μετανάστευσης θα είναι στην ημερήσια διάταξή μας για καιρό ακόμα. Και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό το θέμα και μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου της διάσκεψης κορυφής είναι το θέμα της ασφάλειας. Στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ασφάλεια είναι μια μεγάλη πρόκληση. Η Ευρώπη και ο κόσμος έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Ζούμε σε μια εντελώς διαφορετική γεωπολιτική κατάσταση σήμερα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα δει τι δουλειά έχει γίνει μέχρι τώρα στο θέμα της εσωτερικής ασφάλειας και κατά τη Λετωνική Προεδρία πρέπει να ξέρετε ότι το Συμβούλιο έκανε πολλά για να ενισχύσει την ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 16 Ιουνίου το Συμβούλιο επιβεβαίωσε και ενέκρινε ε, νέα στρατηγική για την εσωτερική ασφάλεια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το έλαβε υπόψη του Έχουμε προχωρήσει σε πολλά ζητήματα. Έχουμε αυξήσει την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές των χωρών μελών. Και από 1η Ιουλίου η μονάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το περιεχόμενο του διαδικτύου θα αρχίσει τις εργασίες της. Πρέπει όμως να συνεχίσουμε προκειμένου να ελέγχουμε ε, περισσότερο τα εξωτερικά μας σύνορα για την ασφάλεια. Ζητούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επαναλάβει τη στήριξή του και την ε, θέση του προκειμένου να αρχίσει τριμερής διάλογος για την ε, σχετική οδηγία για τη μετανάστευση. Η συνεργασία μας επίσης με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης έχει αρχίσει και θα υποβάλουμε στο Συμβούλιο για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Και μια που βρισκόμαστε στην εξωτερική διάσταση, το Συμβούλιο Κορυφής θα συζητήσει και για την ε, κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας και θα αξιολογηθεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί μετά από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2013, το Δεκέμβριο δηλαδή. Η συζήτηση αυτή θα γίνει βέβαια μέσα σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Οι επισημένε προκλήσεις είναι διαφορετικέ. Είναι πάντως σημαντικό να γνωρίζουμε ότι αρχίζουμε τη UNAFORM Φόρμο που είναι μια νέα δράση της κοινή μας πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια νέα στρατηγική για το Συμβούλιο θα ζητήσει από την ΕΠΑ το εκπρόσωπο να προετοιμάσει μια τέτοια νέα στρατηγική. Θα ζητήσουμε επίσης από την ΕΠΑ το εκπρόσωπο να ηγηθεί των εργασιών προκειμένου να ετοιμαστεί και μια ε, στρατηγική ανακοίνωση. Χρειάζεται συντονισμός και από κοινού δράση για ενημέρωση. Χτες και σήμερα επίσης στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων συνεχίστηκε η συζήτηση προκειμένου να έχουμε μια νέα ανακοίνωση. Οι νέες προκλήσεις δείχνουν ότι χρειάζεται συνεργασία για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τις υβριδικές απειλές. Εκτιμούμε λοιπόν θετικά την απόφαση της 18ης Μαΐου του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων να γίνουν νέες προτάσεις προς αντιμετώπιση των υβριδικών αυτών απειλών και ελπίζουμε μέχρι τα τέλη της χρονιάς να τις έχουμε τις προτάσεις αυτές. Ελπίζουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ζητήσει και κινητοποίηση νέων πόρων. Ως Προεδρία αναμένουμε ότι τα θέματα αυτά θα παραμείνουν στην, Ευρω... στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για αρκετούς μήνες. Ευρωβουλευτές. Η ημερήσια διάταξη της διάσκεψης κορυφής περιλαμβάνει και θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία. Οι οικονομικοί δείκτες δείχνουν ότι η κατάσταση βελτιώνεται 1,8% φαίνεται η ανάπτυξη για φέτος και του χρόνου η ανάκαμψη θα φτάσει στο 2,1%. Τα επίπεδα ανεργίας επίσης μειώνονται. Βλέπουμε θετικά αποτελέσματα και εξαιτίας εξωτερικών παραγόντων αλλά και εξαιτίας της εφαρμογής των πολιτικών μας. Πρέπει να συνεχίσουμε όμως να δουλεύουμε υπέρ της οικονομικής ανάπτυξης και της μακροχρόνιας οικονομικής ανάπτυξης τον κύκλο συντονισμού της οικονομικής μας πολιτικής, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο που μόλις έληξε, οι τρεις προτεραιότητες ήταν η πρόθεση των επενδύσεων και η βελτίωση των οικονομικών μας πολιτικών. Βάσει των προτεραιοτήτων αυτών, κάθε χώρα μέλος έχει κάποιες συστάσεις Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα, λέει ο Μιλήτρια. Πράγματι υπάρχει βόμβο στα ακουστικά. <laughs> Okay ekonomikas pārvaldības jomā viena prezidentūras eh, norisi tā jaunajā pilnveidotajā veidolā. Ήμασταν στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο λοιπόν. Υπήρξε ένα τεχνικό πρόβλημα. Με συγχωρείτε, τώρα είναι εντάξει η διερμηνία από ό,τι φαίνεται. Η λετωνική καμπίνα, μισό λεπτό. Εσύ. Ακούγεται καλά τώρα η μετάφραση. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, Όπω σας είπα ήδη, στον τομέα της οικονομικής διακυβέρνησης, μία από τι προτεραιότητε της Λετωνική προεδρία είναι η επιτυχής εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου υπό τη νέα της βελτιωμένη μορφή. Η ανάλυση αναχώρα δημοσιεύτηκε νωρίτερα και δίνουμε περισσότερη σημασία στις αναχώρα συστάσεις. Πρόκειται για την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Μεταρρυθμίσεις οι οποίες είναι αναγκαίες προκειμένου να βελτιωθεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και να πετύχουμε την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η Λετωνική Προεδρία λοιπόν έθεσε τις σωστές βάσεις για συζητήσεις όσον αφορά τις διαρθρωτικές επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις. Μπήκανε οι βάσεις για μακροχρόνια οικονομική ανάπτυξη και θα σας δώσω διάφορα παραδείγματα. Πρώτον, σε ένα χρόνο ρεκόρ μπορέσαμε να συμφωνήσουμε για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω από βάθος καρδίας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έργο τους, που ελπίζουμε θα οδηγήσει σε θετική ψήφο σήμερα. Δεύτερον, το Συμβούλιο το εξάμεινο αυτό έδωσε ιδιαίτερη σημασία στη χρησιμοποίηση των ε, θετικών από την ενία αγορά, προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια που υπάρχουν στην ψηφιακή, για παράδειγμα, ενιαία αγορά. Είμαστε σε ψηφιακή εποχή που σημαίνει ότι αυτή μπορεί να μας βοηθήσει για να μειωθεί η ανεργία και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά μας. Η ψηφιακή τεχνολογία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην καινοτομία και την ανάπτυξη και δεν είναι μόνο οι υπουργοί που το λένε αυτό, Πρέπει να λάβουμε υπόψη μα συνεπώ τη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκή Επιτροπής και το Συμβούλιο δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά τα θέματα. Όχι μόνο για να αρθούν τα εμπόδια από την ενιαία ψηφιακή αγορά. Ελπίζουμε το Συμβούλιο να δώσει νέα όθηση τώρα, η διάσκεψη κορυφή δηλαδή, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νομικές πράξεις που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί η ψηφιακή αγορά. Η Λετωνική Προεδρία κάνει ό,τι μπορεί για να επιτευχθεί πρόοδος επίσης όσον αφορά τον κανονισμό της προστασίας δεδομένων, τηλεπικοινωνιών και ε, ασφάλεια της πληροφορίας. Το Συμβούλιο θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης επίσης. Έχουμε επίσης τώρα πολύ πρόσφατα την έκθεση των πέντε Προέδρων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα έχει μια πρώτη συζήτηση τώρα για αυτό το θέμα και κατά διάρκεια της Προεδρίας του Λουξεμβούργου θα συνεχιστεί το έργο για τα όσα αναφέρονται στην έκθεση αυτή. Η έκθεση μεταξύ άλλων κάνει διάφορες συστάσεις για το πώς να διαχειριστούμε καλύτερα την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, και αύριο οι επικεφαλείς κρατών και κυβερνήσεων θα τα συζητήσουν. Δεν θα ήθελα εδώ όπως καταλαβαίνετε να προκαταλάβω το τι θα συζητήσουν εκείνοι αύριο. Κατά τη γνώμη μου όμως θα υπάρξουν πολλές καλές ιδέες προκειμένου η Οικονομική και Νομισματική Ένωση να γίνει περισσότερο βιώσιμη, πιο ισχυρή και θέλω να υπογραμμίσω επίσης ότι πρέπει να γίνουν πολλά για να πετύχουμε τη σύγκληση. Οι διαφορές μεταξύ των κρατών της Ευρωζώνης μπορούν να αποτελέσουν μια απειλή για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η μέληση διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι γεμάτη από επίκαιρα και σημαντικά θέματα, αλλά είμαι εδώ για να ακούσω τις απόψεις σας, τα σχόλιά σας και προβλέπω σε ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Ευχαριστώ την Προεδρία του Συμβουλίου και τώρα το λόγο θα πάρει ο πρώτος Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Φραντ Τίμερμανς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύρια Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι. Όταν ο πρόεδρος Γιούνκερ αναφέρθηκε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 15 Ιουλίου του προηγούμενου έτους, είπε ότι η πρώτη αποστολή είναι να ξαναδημιουργήσει γέφυρε στην Ευρώπη. Το να φτιάξουμε γέφυρες όμως στην Ευρώπη και πέραν της Ευρώπης είναι ένα πραγματικά ευρωπαϊκό εγχείρημα. Γι' αυτό το λόγο ο κύριος Γιούνκερ δεν είναι παρόν σήμερα μαζί σας. Θα ήθελε να είναι μαζί σας, αλλά προσπαθεί να δημιουργήσει γέφυρες με την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο έχουμε πράξει όλους τους τελευταίους μήνες, τις τελευταίες μέρες με την Ελλάδα είναι η δημιουργία γεφυρών. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι δημιουργημένη για να αποκλείει αλλά για να περιλαμβάνει τα μέλη της. Πρέπει να είναι μια ένωση η οποία θα βασίζεται στην κατανόηση και τον αμοιβαίο σεβασμό. Δεν είναι πάντα εύκολο. Δεν είναι πάντα ένας μακρύς ήρεμος ποταμός, όπως λένε οι λογοτέχνες. Αλλά ο καθένας θα πρέπει να βάλει το πετραδάκι για να δημιουργηθούν αυτά τα γεφύρια. Πρέπει να βρούμε μια συμφωνία <clears throat> αυτή τη βδομάδα σε σχέση με το θέμα της Ελλάδος. Ο χρόνος μας πιέζει. Θα πρέπει να προχωρήσουμε κατευθείαν προς την επίτευξη του στόχου αυτού. Δεν υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω χρονικής παράτασης. Υπάρχει μια απέτηση να δοθούν απαντήσεις στις, στα αιτήματα των Ελλήνων οι οποίοι υποφέρουν και προς αυτούς η στρέφεται η σκέψη της Κομισιόν και του Προέδρου Ιούνκερ. Εργαζόμαστε για να τους βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν την ανεργία, την επισφάλεια στα κοινωνικά θέματα, να οικοδομήσουν το μέλλον της επιστερεών βάσεων. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει όλοι να επομιστούμε τις ευθύνες μας. Και η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρωομάδα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αλλά και το Κοινοβούλιο, η Κομισιόν. Όλοι μας θα πρέπει να δεσμευτούμε ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε στην Ελλάδα μια νέα εκκίνηση για την απασχόληση, την οικονομική μεγέθυνση και τις επενδύσεις χάρη στις μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να επιφέρει αλλά και χάρη στην αρρωγή των ευρωπαϊκών θεσμών. Από τη στιγμή που θα πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις και θα υπάρξει μια συμφωνία, η Κομισιόν είναι έτοιμη να κινητοποιήσει ή μάλλον να επανακινητοποιήσει την εκταμείευση 35 δισεκατομμυρίων ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό για να υποστηρίξει την Ελλάδα. Ο πρόεδρος Γιούγκερ θα προτείνει λύσεις για να διευκολυνθεί η απορρόφηση των διαρθωτικών πόρων και να ενισχυθούν οι ευρωπαϊκές επενδύσεις και να κινητοποιήσει με προχρηματοδότηση σημαντικά ποσά για να ξεκινήσουν επενδύσεις στην πραγματική οικονομία της Ελλάδας. Το τέλος όμως των κοινών προσπαθειών θα μπορέσουμε να βρούμε μια συμφωνία που να είναι αποδεκτή για όλους. Έχουμε κάθε εμπιστοσύνη ότι αυτό θα μπορέσει να γίνει μετά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της αυριανής και μεθαυριανής μέρας. Το να χτίσουμε γέφυρες είναι και πάλι αυτό το οποίο θα πρέπει να είναι η... ο στόχος των προσπαθειών μας τις επόμενες μέρες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Για το θέμα τώρα της μετανάστευσης, το οποίο αναφέρθηκε το Συμβούλιο. Αν υπάρχει ένας χώρος στον οποίο μπορεί να εκφραστεί η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, είναι το θέμα της μετανάστευσης. Ήμουν παρόν χθε στο αρμόδιο Συμβούλιο. Ορισμένε φορές εκπλήσεται κανείς με την ευκολία με την οποία ορισμένα κράτη-μέλη ζητούν την αλληλεγγύη και στη συνέχεια σιωπούν όταν πρέπει και αυτά να δείξουν αλληλεγγύη προς τους άλλους. Όλοι συμφωνούμε για το γεγονός ότι είναι κατεπήγον να δώσουμε μια απάντηση στην ανθρωπιστική και μεταναστευτική κρίση που αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες μας. Πρέπει να το κάνουμε με τον με τον άλλο τρόπο. Όλοι μας αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα και θα το αντιμετωπίσουμε αργά ή γρήγορα. Αλλά του, του λεχθέντος. Το κατεπήγον τώρα είναι να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για το πρακτέο, ώστε η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη να μην είναι ένα κενό γράμμα ή μονάχα ένα δάκρυ το οποίο ε, φεύγει από τα μάτια μας σε κάθε κρίση χωρίς όμως η Ευρώπη να προχωράει. Τα λεπτά σιγής κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν θα πρέπει να ακολουθούνται από σιωπή από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όταν από αυτό περιμένουμε όλοι να δώσει απαντήσεις. Αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει να πράξουμε είναι αυτό. Να απλώσουμε το χέρι μας σε αυτούς τους δυστυχισμένους που με κίνδυνο της ζωής τους φεύγουν από τη χώρα τους θύματα συγκρούσεων, πολέμων για να βρουν μια διεθνή προστασία για την οποία έχουν κάθε δικαίωμα να την διεκδικήσουν είναι θέμα σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Θα πρέπει επίσης να δείξουμε με αυτό τρόπο την αλληλεγγύη μας προς τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν μια πολύ μεγάλη μεταναστευτική πίεση. Η Ιταλία και η Ελλάδα συγκεκριμένα σήμερα. Αύριο μπορεί να είναι και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε όλες τις περιπτώσεις χρειάζονται μηχανισμοί αλληλεγγύης. Τώρα πρέπει να θέσουμε σε εφαρμογή τους μηχανισμούς αυτούς με το να δράσουμε από κοινού και όχι ημέν κατά τον δε. Σήμερα, όχι αύριο. Πεθαίνουν ακόμα άνθρωποι κάθε μέρα στη Μεσόγειο. Ας είμαστε σαφείς. Δεν μιλάμε για ποσοστώσεις όταν πρόκειται για ανθρώπινα όντα. Αυτό είναι μια παρεξήγηση. Μιλάμε για μια κλίδα ανακατανομής, αλλά δεν έχουμε σαν στόχο να θέσουμε σε ό,τι αφορά το δικαίωμα για παροχή ασύλου. Όλοι μας έχουμε την υποχρέωση αλληλεγγύης. Ο πρώτος Γιούνκερ θα υποστηρίξει λοιπόν στεναρά τις προτάσεις της Κομισιόν σε σχέση με την επανεγκατάσταση και την μεταφορά των ετούντων ασύλου, γιατί αυτές οι προτάσεις είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν μια σωστή ισορροπία μεταξύ της αλληλεγγύης και της ευθύνη των κρατών μέλων. Κάνα κράτος μέλος δεν μας έχει προτείνει κάτι καλύτερο. Είπαμε πολλές φορές ότι θέλουμε μια λύση από τα κράτη-μέλη, τα οποία όμως δεν μας έχουν δώσει καμιά αναλλακτική λύση. Η κατανομή λοιπόν, επαναλαμβάνω, μεταξύ κρατών μερών πρέπει να γίνεται επί τη βάση μιας αποτελεσματικής κλίδας. Μας έδειξε η εμπειρία ότι δεν δουλεύουν μονάχα οι εθελοντικές λύσεις στον τομέα αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να συμφωνήσουμε μέχρι το τέλος του Ιουλίου σε σχέση με τους πρακτικούς τρόπους με τους οποίους θα γίνει αυτή η αλληλέγγυα και η ισοδίκια κατανομή μεταξύ των κρατών μελών ώστε να μπορέσουν το ταχύτερο δυνατό να υλοποιηθούν αυτά τα μέτρα. Το κόστος της αδράνειας μας σήμερα θα είναι εξαιρετικά βαρύ και για τους μετανάστες αλλά και για την Ευρώπη. Μια Ευρώπη όπου πρέπει να υπάρξει αλληλεγγύη, πρέπει να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση της αλληλεγγύης, το να μείνουμε χωρίς δράση θα είναι μια άρνηση των αξιών επί των οποίων είναι οικοδομημένη η Ευρωπαϊκή Ένωση και προς τις οποίες είμαστε προσιλωμένοι. Ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν χώρες που έχουν opt-in, άλλες χώρες έχουν opt-out, αυτοεξαιρέσεις, αλλά η Ευρώπη είναι πράγματι αξιόπιστη μόνο όταν αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη και όταν δρά ενωμένη και αλληλεγγύα. Εγώ χαίρομαι για το γεγονός που η Ιρλανδία, η Νορβηγία, η Ελβετία και το Λίχτενστάιν έχουν δηλώσει ότι είναι έτοιμες να συν, ε, συμβάλλουν σε αυτό το μηχανισμό επανεγκατάστασης. Προκαλούμε και άλλες χώρες να εμπνευστούν από αυτό το παράδειγμα. Πρέπει να βοηθήσουμε λοιπόν αυτούς που έχουν ανάγκη διεθνού προστασία, αλλά συγχρόνω θα πρέπει να είμαστε στεναροί έναντι αυτών που δεν έχουν κανένα λόγο να παραμείνουν στην Ευρώπη και δεν έχουν κανένα λόγο να ζητούν διεθνή προστασία. Γι' αυτό έχουμε παρουσιάσει προτάσεις για να ενισχύσουμε τι ε, μα μας σε ό,τι αφορά την επανεισδοχή και την επιστροφή των μεταναστών. Γιατί η υποστήριξη στις πολιτικές υπέρ της παροχής ασύλου μειώνεται στον πληθυσμό όταν πιστεύουν πολλοί ότι είναι πολλά άτομα που εκμεταλλεύονται αυτή την πολιτική ενώ δεν έχουν δικαίωμα σύλλου. Πρέπει λοιπόν να συνδυάσουμε και τα δύο. Ο στόχος μας δεν είναι να αντιμετωπίσουμε τα συμπτώματα της κρίσης και μόνο. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με τις χώρες διέλευσης και προέλευσης για να αντιμετωπίσουμε τις ρίζες της κρίσης. Την αιτία την ξέρουμε. Η αστάθεια, ο πόλεμος, η ένδια στη Λιβύη, στη Συρία, στο Ιράκ και σε ένα μεγάλο μέρος της Αφρικής και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δημιουργήσουμε γέφυρες και να έχουμε περισσότερη κοινή ευθύνη, περισσότερη συνεργασία με τους Αφρικανούς εταίρους μας. Με κάθε τίμημα πρέπει τα κράτη-μέλη να αυξήσουν την αναπτυξιακή τους βοήθεια. Αυτό είναι απαραίτητο. Χρειαζόμαστε να πετύχουμε όλοι το στόχο του 0,7% σήμερα, όχι αύριο, όχι σε χρόνια από σήμερα. Για τα θέματα άμυνας. Τη στιγμή που η Ουκρανία και η Συρία, η Μέση Ανατολή και η Βόρεια Αφρική είναι όλο και πιο αυστατής και ευάλωτη, θα πρέπει να είμαστε αφελείς για να νομίζουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να είναι μονάχα μία ήπια δύναμη. Δεν μπορεί να υπάρξει ήπια δύναμη σε βιώσιμο επίπεδο χωρίς και σκληρή δύναμη, χωρίς ικανότητα άμυνας. Είναι και αυτό ένα θέμα αξιοπιστία. Δεν σημαίνει ότι από τη μια μέρα στην άλλη πρέπει να προχωρήσουμε προ ένα ευρωπαϊκό στρατό. Αυτό είναι ένα παλιό εγχείρημα, ένα εγχείρημα το οποίο έχει μακροχρόνιο χαρακτήρα. Ούτε πρόκειται να κάνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα αντίπαλο του ΝΑΤΟ. Δεν είμαστε ανταγωνιστέ, είμαστε εταίροι. Θα πρέπει από κοινού να εργαστούμε και να βρισκόμαστε στο ίδιο μήκο κύματο. Για τον αμυντικό τομέα αυτό το οποίο χρειάζεται μια ενισχυμένη συνεργασία όπως προβλέπει και η Συνθήκη της Να κάνουμε περισσότερα από κοινού για να επιτύχουμε περισσότερα από ό,τι μπορούμε να πετύχουμε με μεμονωμένες και μόνο εθνικές ενέργειες. Σήμερα στην Ευρώπη πάνω από 80% των επενδύσεων σε εξοπλισμούς γίνονται σε εθνικό επίπεδο. Ακόμα και για λόγους μονάχα οικονομίας, για λόγους προϋπολογισμού, θα πρέπει να δημιουργήσουμε γέφυρες συνεργασίας στις αγορές εξοπλισμού, στην έρευνα και την ανάπτυξη για να μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας και να ανταποκριθούμε στις κοινέ προκλήσεις. Εν τέλει θα πρέπει να έχουμε γέφυρες και προς το μέλλον και να συμπληρώσουμε την Οικονομική και Νομισματική Ένωση διατηρώντας την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς. Μας έδειξε η κρίση ότι το ευρώ μας προστατεύει, μας δίνει νομισματική σταθερότητα. Χωρίς το ευρώ θα είχαμε περάσει πολύ δύσκολες και δυσάρεστες στιγμές θα είχαμε δει έξαρση των εθνικών οργανισμών. Αλλά η προστασία του ευρώ δεν έρχεται από τον ουρανό. Συνδέεται με την αξιοπιστία μας όταν θέτουμε ε, σε ισχύ πολιτικές οι οποίες βασίζονται σε εξισορροπημένη ε, οικονομική ανάπτυξη, σε μια κοινωνική οικονομία της αγοράς που υποστηρίζει και την κοινωνική ε, ανάπτυξη και την ευμάρεια των πολιτών. Αυτή ακριβώς και είναι η στόχη αυτής της ε, μελέτης και από ό,τι καταλαβαίνω σωστά τα λέει η μετάφραση. Αυτός είναι και ο στόχος της έκθεσης των πέντε πρόεδρων διότι ο πρόεδρος Γιούγκερ θέλησε να συμμετάσχει σε αυτό το εγχείρημα και ο πρόεδρος Σούλτς. Υπάρχει ένα οδικός χάρτης για τη συμπληρώση οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Είναι μια φιλόδοξη αλλά και πραγματιστική προσέγγιση και κάποιες από τις πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται μπορούν ήδη σήμερα να εφαρμοστούν. Τα πρώτα μέτρα θα πρέπει να ξεκινήσουν από τους θεσμούς από την 1η Ιουλίου 2015. Άλλο χρόνο, αλλά κινούνται προς μια σαφή κατάσταση που είναι ουσιαστική για τους οικονομικούς φορείς και τους πολίτες και για την εμπιστοσύνη στο ενιαίο νόμισμα. Η πρώτη φάση που θα πρέπει να υπάρξει εμβάθυνση, ξεκινά ήδη από σήμερα μέχρι τον Ιούνιο του 2017. Βασίζεται στα υπάρχοντα εργαλεία και τις συνθήκες που ήδη είναι ενισχύ για να υπάρξει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, μεγαλύτερη σύγκληση, πιο υπεύθυνη πολιτική σε δημοσιονομικά επίπεδα, να ενισχυθεί η αλληλεγγύη και να ενισχυθεί και η υπευθυνότητα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Η δεύτερη φάση, σε δημοκρατικό επίπεδο, η δεύτερη φάση θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε σε δράσεις μεγαλύτερης εμβέλειας για να μπορέσει η διαδικασία σύγκλησης να γίνει πιο περιοριστική και να δημιουργηθεί και ένας προϋπολογισμός για τη ζώνη του ευρώ. Η τελευταία φάση θα οδηγήσει σε ένα μέλλον σταθερό και ευμαρές για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν μπει στη ζώνη του ευρώ και θα είναι και ελκυστική και για τις άλλες χώρες. Με σταδιακό τρόπο λοιπόν και μεγαλύτερο τρόπο θέλουμε να δημιουργήσουμε μια οικονομική ένωση, μια ένωση κεφαλαίων, μια ένωση προπολογισμού και εν τέλει μια πολιτική ένωση. Αυτό δεν είναι αυτός σκοπός, αλλά ένας τρόπος να αντιμετωπίσουμε τα αιτήματα των πολιτών και τις προσδοκίες τους και να προετοιμάσουμε την Ευρώπη για τις μελλοντικές παγκόσμιες προκλήσεις. Η Ευρώπη είναι κάτι περισσότερο από μια ενιαία αγορά, μια οικονομική και νομισματική ένωση. Είναι ένα τεράστιο εγχείρημα για τους πολίτες αλλά και πέραν των πολιτών τους. Πρόεδρε, θα τελειώσω στη μητρική μου γλώσσα. Σήμερα στην Ολλανδία έχουμε μια μουσική εκδήλωση πολύ αγαπητή από τον κόσμο. Θέλω λοιπόν να σας πω κάποια λόγια από αυτά που συνηθίζουμε να λέμε αυτή τη μέρα τα οποία αντικατοπτρίζουν πολύ καλά και το πνεύμα των ημερών. Όλοι ανήκουμε στον κόσμο και ο κόσμος είναι όλοι εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος του ΕΛΚΑ έχει τώρα το λόγο ο κύριος Βέμπερ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε τη Κομισιόν, κυρία Πρόεδρε του Συμβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να σταθώ σε δύο μονάχα σημεία τα οποία έχουν συζητηθεί στο Συμβούλιο και θα αντιμετωπιστούν και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι το θέμα της Ευρωζώνης και του κοινού νομίσματος και της αντιμετώπισης της Ελλάδος. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θέλει η Ελλάδα να παραμείνει στη ζώνη του ευρώ. Βλέπουμε ότι είναι δύσκολη η κατάσταση σήμερα, δεν έχουμε καταλήξει ακόμα σε μια κοινή απόφαση. Γι' αυτό υποστηρίζουμε, υποστηρίζουμε πλήρως τον ε, Jean-Claude Juncker για τις προσπάθειες που καταβάλει. Θέλουμε να τονίσουμε ότι έχουμε αντιμετωπίσει την κρίση αυτή ως Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από την χρηματοπιστωτική κρίση έχει θίξει και άλλες χώρες, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιρλανδία και την Κύπρο, αλλά οι χώρες αυτές έχουν καταφέρει να ξανασταθούν στα πόδια τους μετά από τα προγράμματα που επιβλήθηκαν. Παραμένει ως μεγάλο ερωτηματικό τώρα αυτή η εβδομάδα η Ελλάδα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Έχουμε κάποια αίσθηση ματέωσης, γιατί έχει χαθεί πάρα πολλής χώρος, χρόνος, έχουν γίνει συζητήσεις επί πολλούς μήνες σε τεχνικό επίπεδο, δεν έχουμε καταλήξει πουθενά γιατί η νέα ελληνική κυβέρνηση δεν ήταν σε θέση να καταθέσει αξιόπιστες προτάσεις. Μόνο τη Δευτέρα έγινε δυνατόν να υπάρχει τουλάχιστον ένα κείμενο από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης και μετά από πέντε μήνες που είχε η Ελλάδα αυτή την κομμουνιστική κυβέρνηση το ερώτημα είναι τι έχει επιτύχει αυτή η κυβέρνηση για τη χώρα της. Είχαν πάρει μια χώρα η οποία είπαν ότι ήταν κατεστραμμένη και θέλαν να την ανοικοδομήσουν. Ελπίζαμε λοιπόν από τον Ιανουάριο ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένα πλεόνασμα για το 2015 και τώρα έχει εξαφανιστεί αυτό το πλεόνασμα, έχει και πάλι έλλειμμα ο προϋπολογισμός και στο τέλος του μηνός δεν θα μπορέσουν να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις. Μετά από τόσο δύσκολα χρόνια είχαμε ήδη τον Ιανουάριο μια μικρή οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα. Τώρα έχουμε μια σοβαρή ύφεση. Κανείς δεν θέλει κάτι τέτοιο στην Ευρώπη. Έχουμε τράπεζες οι οποίες ήταν σταθερές και τώρα βρίσκονται ενώπιον ενός bank run, μιας μαζικής ε, απόστησης καταθέσεων, γιατί δεν εμπιστεύεται κανείς από τους πολίτες στην Ελλάδα το σύστημα. Και είναι καιρός επιτέλους οι πλούσιοι να πληρώσουν στην ε, Ελλάδα. Είχε δοθεί αυτή η υπόσχεση πριν από πες ότι θα πληρώσουν επιτέλους οι πλούσιοι στην Ελλάδα. Αλλά μια κομμουνιστική κυβέρνηση γιατί δεν το έχει φέρει αυτό σε πέρας. Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σε ένα τέτοιο απολογισμό μετά από πέντε μήνες, πέντε μήνες κυβέρνησης Τσίπρα. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε τις προσπάθειες, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Το ΕΛΚ θεωρεί ότι η αιρεσιμότητα είναι πάρα πολύ σημαντική. Η Ελλάδα χρειάζεται ένα σχέδιο με το οποίο θα βγει από αυτήν την αρνητική ε, πορεία στην οποία έχει εγκλωβιστεί. Γι' αυτό επιμένουμε για ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι αποτέλεσμα συμφωνίας των δανειστών και της Ελλάδος, αλλά το οποίο θα δώσει επιτέλους προοπτικές στην Ελλάδα. Και τονίζω ότι η μπάλα βρίσκεται στο ελληνικό γήπεδο, στο ελληνικό κομμάτι του γήπεδου. Πρέπει από την Ελλάδα να προέρθουν οι λύσεις και πρέπει να υπάρξει μια πλειοψηφία του ε, ελληνικού κοινοβουλίου, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσει ο Τσίπρας και ο Βαρουφάκης να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των ευρωπαϊκών λαών. Βλέπουμε ότι υπάρχει πραγματικά μεγάλη απογοήτευση από εμά για την δράση της ελληνικής κυβέρνησης. Παρ' αυτά θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια και θα υποστηρίξουμε όλες τις ενέργειες οι οποίες οδηγούν να κρατήσουν την Ελλάδα στο ευρώ. Δεν φταίνε οι άνθρωποι στην Ελλάδα, φταίει η κυβέρνηση. Υπήρξαν χιλιάδες που κατέβηκαν στους δρόμους της Αθήνας τονίζοντα ότι θέλουν να μείνουν στη ζώνη του ευρώ και θέλουν τη βοήθεια της Ευρώπης και εμείς είμαστε στον πλευρό αυτών των ανθρώπων. Θέλω δύο σημεία ακόμα να τονίσω και γιατί αναφερθήκαμε στην προβληματική της μετανάστευσης. Χρειαζόμαστε νόμιμους τρόπους μετανάστευσης προς την Ευρώπη για αυτούς οι οποίοι χρειάζονται την υποστήριξή μας. Η πρόταση της Κομισιόν για την επανεγκατάσταση των σύρων προσφύγων είναι μια θετική πρόταση, μια πρόταση που κανείς δεν μπορεί να απορρίψει, γι' αυτό υποστηρίζουμε απόλυτα την Κομισιόν, του ζητούμε να συνεχίσουν τις προσπάθειες και πρέπει τα κράτη-μέλη να δεσμευτούν να δώσουν βοήθεια στους Σύριους πρόσφυγες όπως καθορίζονται από τον ΟΗΕ. Είναι απαραίτητο λοιπόν να αντιμετωπίσουμε παράλληλα και την κατάχρηση ε, των αιτήσεων ασύλου. Τα δύο τρίτα αυτών των αιτήσεων που έγιναν στην Ευρώπη απορρίφθηκαν. Θα πρέπει να είμαστε σαφείς ότι η Ευρώπη θα πρέπει να εξασφαλίσει τα εξωτερικά της σύνορα. Είμαστε στα ε, στα πλαίσια μιας ε, υπήρου που δεν μπορεί να δέχεται άτομα τα οποία δεν έχουν κανένα νόμιμο λόγο εισόδου μέσα στην Ευρώπη. Και επίσης από, τους, από τις χώρες που είναι υποψήφιες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι η Σερβία, δεν μπορούμε να δεχόμαστε ε, άτομα που ζητούν ε, άσυλο. Επίσης ζητούμε από την Τουρκία να δεχθεί αυτούς οι οποίοι επιστρέφονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητούμε επίσης από τον Αντιπρόεδρο της ε, Επιτροπής να συνεχίσει όπως ε, είπε τις συζητήσεις με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης στην Αφρικανική Ήπειρο. Χρειαζόμαστε μια εξισορροπημένη πρόταση. Βοήθεια από τη μία πλευρά χρειαζόμαστε να ε, διαφοροποιηθούμε από τις ακραίες δυνάμεις στην Ευρώπη που είναι κατά κάθε μετανάστευση, αλλά συγχρόνω να εξασφαλίσουμε και την σταθερότητα και την ασφάλεια τη Ευρωπαϊκή Υπήρου. Ευχαριστώ. Εξ ονόματο ε, του Προοδευτική ε, Συμμαχία ε, Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, το λόγο έχει ο Πρόεδρο Πιτέλα. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ την Υφυπουργό για την εισήγηση που μας έκανε. Ωστόσο, πρέπει να δούμε, ελπίζαμε, να δούμε την τελική κατάληξη της λικής υπόθεσης. Ε, γι' αυτό ακόμα περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει συμφωνία. Το Φεβρουάριο ακούγαμε τα ίδια, τον Απρίλιο το ίδιο. Φαίνηκε να φτάνουμε επιτέλους σε συμφωνία. Ε, πιστεύω πως αυτή θα είναι η καλή φορά. Αλλά εξακολουθώ να ακούω επικρίσεις κάποιοι εκπρόσωποι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, κάποιες προσωπικότητες της ε, Ευρωπαϊκής Δεξιάς και λυπούμε που ένας άνθρωπος που εκτιμώ πολύ όπως ο συνάδελφος ε, Βέμπερ ε, λέει ακόμα σήμερα στις 3 η ώρα πως η, Ευρωπαϊκή, ελληνική προ... κυβέρνηση πρέπει να κάνει προτάσεις. Μα η συμφωνία υπάρχει, είναι επιτάπητος και έχει επιτευχθεί κυρίως χάρη στην προσπάθεια του Προέδρου Γιούνκερ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, στην οποία θα πρέπει να ε, ευχαριστήσουμε και η οποία φρόντισε για μια ισορροπία. Μα τι πρέπει ακόμα να περιμένουμε. Ε, ε θα πέσουμε στη γελιότητα για κάποια ποσοστά ΦΠΑ, ε, εστιατόρια, θα τεθεί σε κίνδυνο η ακαιρεότητα της Ευρωζώνης και του ευρώ και το μέλλον της Ευρώπης. Μα τι παιχνίδι είναι αυτό που παίζουμε. Αν κανένα θέλει να ταπεινώσει τον ελληνικό λαό κάνει λάθο, Οι κυβερνήσει. και εμεί δεν είμαστε η κυβέρνηση Τσίπρα, οι κυβερνήσει αλλάζουν με την ψήφα των πολιτών. Και αυτή τη στιγμή δεν αμφισβητείται η κυβέρνηση Τσίπρα, ούτε και οι κρίσεις για την κυβέρνηση Τσίπρα. Είναι υποσυζήτηση η διάσωση του ελληνικού λαού και η διάσωση της ακεραιότητας της Ευρωζώνης. Το να παρατείνονται τεχνικές συζητήσεις... Ε, επιφέρει το κίνδυνο και αποκαλύπτει το κίνδυνο μιας ε, γραφειοκρατική Ευρώπη χωρίς όραμα και για τη μετανάστευση. Και εγώ ευχαριστώ τον Πρόεδρο Τίμερμανς που έκανε μια στεναρή συμπαγή ε, ομιλία με όραμα. Αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο και στο εσωτερικό του Συμβουλίου και πρέπει να το πω αυτό πολύ ειλικρινά και προ μεγάλη μου θλίψη. Υπάρχουν από την μια πλευρά χώρε όπω η Ιταλία που δεσμεύονται για να κάνουν ό,τι μπορούν για να σώσουν την ανθρώπινη ζωή στη Μεσόγειο ε, και υπάρχουν από την άλλη κάποιε κυβερνήσει όπω αυτή τη Ουγγαρία που υψώνουν ε, τύχη ε, μπροστά στους μετανάστες. Πραγματικά, τι θλίψε Μια χώρα όπως η Ουγγαρία, η οποία ύψωσε το σιδηρούν, μάλλον που έζησε το σιδηρούν παραπέδασμα, να ε, κατασκευάζει νέα ατύχη απέναντι στους μετανάστες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δίκιο. Εν μέρη φαίνεται να γίνεται αποδεκτή η πρόταση από το κράτη-μέλη. 40.000 ε, μετανάστες, δημιουργία hot spots. Και εντάξει, αλλά δεν αρκούν όλα αυτά. Κατανοώ τη διπλωματία, αλλά δεν μπορούμε όλα να τα περιορίζουμε σε, ένα γλωσσικό, σε μια γλωσσική και αμφίσιμη άσκηση. Λέει ότι ορισμένα κράτη είναι υπέρ της αλληλεγγύης, αλλά είναι κατά των υποχρεωτικών μηχανισμών. Μα τι σημαίνει αυτό. Κάποιος πρέπει να με εξηγήσει τι σημαίνει αυτό. Ναι ε, υποχρεωτικοί μηχανισμοί γιόκ. Μα τι θα πει. Εξηγήστε το μου, εξηγήσατε μου τι σημαίνει συγκεκριμένα. Και ε, ε, μπρο σε ένα τόσο ουσιαστικό θέμα τι κάνουμε. Ξεφεύγουμε με λόγια κάνουμε τους έξυπνους μόνο με τα λόγια, αντί να μπούμε στην ουσία και να δείξουμε ότι είμαστε στο ύψος μιας περίστασης, να είμαστε ηγέτες της Ευρώπης. Αν δεν είμαστε ηγέτες, και το λέω στις κυβερνήσεις, γιατί φοβούμαστε, γιατί φοβόμαστε για τις ε, λαϊκιστικές ε, ε, εξάρσεις. Αυτά όλα είναι αποτέλεσμα καρπός της έλλειψης ε, δύναμης. Αν μια, το ένα κράτος ε, εναντιώνεται στο άλλο, αν αρχίζουμε και τσακωνόμαστε μεταξύ μας, αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχει ένα ευρωπαϊκό όραμα. Γι' αυτό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κάθε δικαίωμα να υψώσει τη φωνή του. Αυτό, αυτή είναι στην αίθουσα όπου έχουμε και κάποιες μειοψηφίες των οποίων δεν συμμερίζομαι την άποψη. Σε αυτή την αίθουσα λοιπόν και σε αυτό το θέμα ανέκαθεν ναι, εκφράζαμε ισχυρές θέσεις και θέλω να τις, αυτές να επαναλάβω και να υπογραμμίσω μέσω της παρέμβασής μου. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος της ομάδας των συντηρητικών μεταρρυθμιστών της Ευρώπης έχει το λόγο ο κύριος Καμάλ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ τη Λετωνική Προεδρία. Είπατε ότι είναι η τελευταία ολομέλεια που βρίσκεστε εδώ. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα. Όποιο και είναι το πρόβλημα, οι λύσει που προτείνονται είναι περισσότερε ρυθμίσει και περισσότερη Ευρώπη. Εμεί όμω είμαστε κατά τη γραφειοκρατίας, είμαστε υπέρ της δημιουργίας απασχόλησης. Και ελπίζουμε αυτά τα πράγματα να συζητιώνται στην Σύνοδο. Η Ελλάδα, η μετανάστευση, αλλά με λύση όχι περισσότερη γραφειοκρατία, όχι περισσότερη Ευρώπη, όχι. Κάτι που θα βοηθήσει την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, να μην έχουμε μια νέα κρίση. Εμείς, ε, αντί να δώσουμε ένα πραγματικό φάρμακο, βάζουμε τσιρότα μόνο. Ε, δεν φτάνουν αυτά. Μέχρι την επόμενη κρίση που θα έχουμε. Και πάλι το ίδιο θα κάνουμε πάλι τσιρότο, μέχρι την επόμενη μεγάλη κρίση και ούτω καθεξής. Μα μέχρι πότε, πόσο θα μας πάρει μέχρι να ξαναβρεθούμε εδώ και να ξεζητάμε τα ίδια και τα ίδια. Πόσο πια τσιρότο θα κολλήσει η Ευρωζώνη. Κάποια στιγμή θα τελειώσει και αυτό. Λένε οι χώρες του ευρώ ότι μπορούν να κρατήσουν την Ελλάδα μέσα στην Ευρωζώνη. Δεν είναι όμως ειλικρινείς με τους πολίτες τους τα χρήματα δεν πάνε από τους πλούσιους στους στοχούς. Και η ελληνική κυβέρνηση έχει και το δικό της ρόλο να παίξει και να αναλάβει τις δικές της ευθύνες όπως είπαν και άλλοι εδώ. Μα πρέπει να σταματήσει πια αυτό. Πρέπει να αρχίσουμε να τηρούμε τους κανόνες όσοι έχουν και όχι να τους παρακάμπτουμε. Δεν μπορούμε να αφήσουμε οποιοδήποτε να μπει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι καλώς πρέπει να έχουμε συγκεκριμένους κανόνες και σίγουρα τους ανθρώπους που κινδυνεύουν στη θάλασσα δεν πρέπει να τους αφήνουμε να πνίγονται, αλλά πρέπει να τηρούμε τους κανόνες, να αποφύγεται αυτή η λαθρέα μεταφορά ανθρώπων στις χώρες μας και όσοι είναι όντως κυνηγημένοι να τους κρατάμε. Αντί όμως για τη συνεργασία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει κάτι άλλο. Αντί για την αλληλεγγύη έχουμε τώρα πόλωση. Αντί να συνεργαζόμαστε, τσακωνόμαστε μεταξύ μας οι χώρες μας. Μας βρεθούμε επιπλέ, επιτέλους σε ένα πνεύμα συνεργασίας μεταξύ μας και να βοηθήσουμε τις χώρες εκεί που υποφέρουν οι άνθρωποι. Και πριν μπουν στο ταξίδι αυτό οι άνθρωποι να ξέρουν αν τους θέλουμε δεν τους θέλουμε. Μην βάλουμε τσιρότο και σε αυτή την κρίση. Ασφάλεια και άμυνα τώρα συνεργασία ή συντονισμός, αλλά όχι συγχώνευση. Η μία χώρα μετά την άλλη, η μία εκλογή μετά την άλλη. Ο κόσμος λέει αυτό που λέει η ομάδα μας, το ECR, ότι η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει, ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργό ο Κάμερον, χρειάζονται μεταρρυθμίσεις. Εμείς δεν πρέπει να το έχουμε σαν ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο που θα παίρνουμε ό,τι δώρο θέλουμε και μας κάνει. Όχι όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Προκλήσεις που έχουμε στα σύνορά μας, προκλήσεις που έχουμε στις χώρες μας, αλλά και εκτός των σύνορων μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος της ε, Συμμαχίας των Δημοκρατών και των Φιλελεύθερων, ο κύριος Φερχόφστατ. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να πω στον κύριο Τίμερμανς ότι νόμιζα πως στο τέλος θα τραγουδούσε, αλλά δεν το έκανε. Αλλά συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπατε για τη μετανάστευση και με τις προτάσεις που υποβάλλατε. Η μόνη μου παρατήρηση λοιπόν είναι ότι θα πρέπει να είστε συνεπείς για όλα αυτά. Τα όσα είπατε είναι αλήθεια, αλλά αυτά που είδαμε τώρα με την Ουγγαρία και ο κύριος Πιτέλο αναφέρθηκε σε αυτό είναι σκάνδαλο από μόνο του. Γιατί είναι έναντι, εναντίον του κοινοτικού κεκτημένου, εναντίον της κοινή προσέγγισης και της προσέγγισης αλληλεγγύης που εσείς υπερασπιστήκατε εδώ στην ε, αίθουσα τούτη. Ελπίζω λοιπόν ότι στο τέλος της δεύτερης σας παρέμβασης και σε επόμενες ε, μέρες η Κομισιόν θα καθαστήσει σαφές ότι τα όσα κάνει ο κ. Ορμπάν είναι ε, κατά των κανόνων της Ευρώπης και ότι δεν μπορούμε να τα δεχτούμε και για τα τείχη που φτιάχνει και για όλα. Λοιπόν, δεύτερη μου παρατήρηση για την Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα βγει κάποια συμφωνία, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να φτάσουμε σε συμφωνία και δεν υπάρχει δεν υπάρχει άλλη διέξοδο γιατί μια έξοδο τη Ελλάδα θα ήταν το χειρότερο για τον ελληνικό λαό. Γιατί πάλι θα χάνανε αγοραστική δύναμη, θα γινόταν υποτίμηση και θα έπρεπε να είναι και, και θα είναι και σίγουρα κακό για την Ευρώπη, για την Ευρωζώνη. Γιατί δείχνει πω το ευρώ δεν είναι σταθερό νόμισμα. Μπορεί κανεί να μπαίνει, όποτε θέλει. Είναι σαν πάρτι. Μπαίνει όταν έχει χρήμα, όταν δεν έχει, φεύγει. Ελπίζω λοιπόν πως θα βγούμε. Βρούμε μια λύση. Αλλά θα είναι διαρκής. Ας είμαστε ειλικρινείς. Μιλάμε για αυτά δις από το δεύτερο πακέτο. Δεν λέμε για λύση τώρα για την Ελλάδα. Μιλάμε πώ θα φύγουν αυτά τα 7 δι του δεύτερου πακέτου και όλοι γνωρίζουμε και όλοι το γράφουν ότι θα πρέπει να συζητηθεί και ένα τρίτο πακέτο, συζητηθεί και ένα τρίτο πακέτο για το μέλλον και ότι θα είναι απαραίτητο να βρεθεί μια βασική λύση για την Ελλάδα διότι αυτή δεν είναι τώρα εδώ λύση μια θεμελιώδης λύση για την Ελλάδα βασίζεται σε δύο στοιχεία αγαπητοί συνάδελφοι. Το πρώτο είναι ότι στην Ελλάδα πρέπει επιπλέον να πάψει το πελατειακό και διαφθαρμένο σύστημα που υπάρχει, ο υπερμεγέθης δημόσιος τομέας, η κλειστή αγορά και, τα... και αυτά δεν έχουν γίνει. Δεν σημαίνει ότι... Ε, λίγα παίρνουμε από τους χαμηλόμισθους, λίγα από τους χαμηλοσυνταξιούχους. Όχι, πρέπει να αλλάξει εκβάθρον το σύστημα που υπάρχει. Και αυτό δεν, δεν συμβαίνει και με αυτή τη συμφωνία που κάνουμε για την ώρα, που συζητιέται, εν περιπτώσει, για την ώρα. Και έπειτα άλλη λύση. Διαχείριση του χρέου στην Ευρώπη. Θα ήταν πολύ καλύτερα αν είχαν ακούσει το Κοινοβούλιο και αν είχαν αρχίσει πριν από τρία χρόνια με εκείνο το Ταμείο διάσωση. Θα είχε λυθεί το πρόβλημα. Και τώρα Τώρα τι έχουμε μπροστά μας, μια χώρα όπως η Ευρώπη που ζητά λεφτά, ε, οι άλλοι λένε όχι εμείς δεν δίνουμε χρήματα γιατί εμείς δεν λάβαμε τα ίδια. Ενώ αν είχαμε φτιάξει το Ταμείο Διάσωσης όλοι θα είχαν πάρει την ίδια βοήθεια. Και αυτό ήταν ο σωστός τρόπος για να ε, λυθεί. Και τέλος για την έκθεση. Εγώ ε, είμαι ευχαριστημένο με αυτή την έκθεση, η ολοκλήρωση τη Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Είμαι ευχαριστημένο με την έκθεση των πέντε Προέδρων. Είναι καλή βάση, δεν είναι πλήρη νομίζω. Για παράδειγμα, το Ταμείο Διάσωση ε, δεν περιλαμβάνεται εκεί. Αλλά είναι μια καλή βάση για να ξεκινήσει κανεί και ελπίζω πω εδώ στο Κοινοβούλιο θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε αυτή την πρόταση του τουλεχθέντο. Να σα πω και κάτι ακόμα, αγαπητοί συνάδελφοι, και το λέω και άμεσα στον κύριο Πιτέλα και στον κύριο Βέμπερ, ότι θα ψηφίσουμε. Σε πέντε ώρες θα ψηφίσουμε για μια έκθεση. Την έκθεση Μπερές. Και είναι λιγότερο φιλόδοξη από το έγγραφο των πέντε προέδρων. Μα τι κάνουμε εδώ πέρα. Αυτό το κοινοβούλιο που ανέκαθεν ήταν ε, ηγετικός ο ρόλος του θα ψηφίσει μία έκθεση χωρίς καν να ασχοληθεί με το θέμα. Εντάξει κύριε Βέμπερ, ξέρουμε πώς πάνε τα πράγματα, κάνατε τη συμφωνιούλα σας, ε, το μειώσατε, είπατε ότι είναι έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας, εντάξει. Έχω δει πολύ καλύτερε εκθέσει από την Περβάνς ε, Μπέρες. γιατί δεν ε, τα βάζω με την Περβάνς Μπέρες; Έχω δει πολύ καλύτερε εκθέσει. Πάντως, πριν από την αρχή της ψηφοφορία, κύριε Πρόεδρε, εγώ θα ζητήσω να παραπευθεί στην Επιτροπή, διότι είναι πραγματικά τρελή και άχρηστη αυτή η έκθεση. Και το λέω όλους τους συναδέλφους, είναι τρελό να ξεκινάμε μια ψηφοφορία για μια έκθεση που έχει ήδη ε, έχει ήδη πεταχτεί στο καλάθι των αχρήστων λόγω μιας καλής πρότασης των πέντε πρόεδρων. Ευχαριστώ για την Γκουε. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Παπαδημούλης. Τη Δευτέρα είδα ανακοινώσεις που θεωρούσαν επιθύρες τη λύση για το ελληνικό πρόβλημα. Η ανακοίνωση του Eurogroup τη θεωρούσε πολύ καλή, η Κομισιόν τη χαιρέτησε ως μια πολύ καλή βάση. Στη Σύνοδο Κορυφής όλοι έλεγαν ότι είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία και ξαφνικά άρχισε η εσωτερική υπονόμευση. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και κάποιες συντηρητικές κυβερνήσεις που αποτελούν μειοψηφία με στην Ευρώπη δείχνουν να μην θέλουν συμφωνία παρότι αυτό είναι το κοινό συμφέρον και της Ελλάδας και της Ευρώπης αλλά αντίθετα θέλουν να την υπονομεύσουν και θέλουν να ταπεινώσουν τον ελληνικό λαό, να αμφισβητήσουν την ανάγκη να σεβόμαστε όχι μόνο τους κανόνες αλλά και τη δημοκρατία. Η ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία και με τις υπηρεσίες της Κομισιόν κατέθεσε μια πρόταση που εξασφαλίζει νοικοκυρεμένα δημόσια οικονομικά με πρωτογενή πλεονάσματα που προωθεί μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, της διαφθοράς, του πελατειακού κράτους, που βάζει τέλος στο έσχος των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων ανθρώπων σε ηλικία 40 και 50 ετών, που οι δικοί σας πολιτικοί φίλοι, κύριε Βέμπερ, εψήφισαν και εφάρμοζαν στην Ελλάδα επί δεκαετίες και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και σας παρακαλώ να αφήσετε τη μισαλοδοξία, Είναι ώρα να συμβάλλουν όλοι στο να υπάρξουν λύσεις για να φύγει η λέξη Brexit από το λεξιλόγιο της ευρωπαϊκής συζήτησης. Για να μπει ο ελληνικός λαός και η Ελλάδα στο δρόμο της ανάπτυξης. Και μη μας κουνάτε το δάχτυλο, κύριοι του Συντηρητικού Κόμματος. Γιατί εφαρμόσατε μαζί με την Τρόικα παραβιάζοντας τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια πολιτική που προκάλεσε κοπές μισθών και συντάξεων 30%, τριπλασίασε την ανεργία, έφερε ύφεση 25% και εκτείναξε το χρέος από το 125% στο 180% του ΑΕΠ. Χρειαζόμαστε νοικοκυρεμένα δημόσια οικονομικά, αλλά και ανάπτυξη και βιώσιμο χρέος. Και αυτό είναι πρόβλημα ευρωπαϊκό πολιτικό και πρέπει να λυθεί με κοινή ευθύνη. Καταθέσαμε προτάσεις, καταθέσαμε ισοδύναμα και τώρα λένε κάτι από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν μας αρέσουν τα ισοδύναμα. Γιατί, γιατί φορολογούμε τους πλούσιους, γιατί φορολογούμε αυτούς που έχουν εισόδημα πάνω από 50.000 ευρώ το χρόνο, για αυτούς που έχουν κέρδη πάνω από 500.000 ευρώ το χρόνο, σε μια χώρα που έχει 1,5 εκατομμύριο ανέργους και που 9 στους 10 ανέργους δεν παίρνουν ούτε ένα ευρώ. Το μήνυμα της πολιτικής μου ομάδας είναι σαφές. Χρειάζεται λύση, επίγει, είναι απολύτως εφικτή, είναι έτοιμη στη βάση αυτών που κατατέθηκαν και θεωρήθηκαν βάση συζήτηση τη Δευτέρα. Κύριε Τίμερμανς, εργαστείτε πάνω σε αυτά. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν είναι υποχρεωτικό να είναι στην καρδιά της Ευρώπης ΕΣΑΗ. E. Η Ευρώπη έχει και τους μηχανισμούς και τους θεσμούς να δώσει απάντηση σε αυτά. Σεβόμενη τη δημοκρατία, η Ελλάδα και η ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη να συμφωνήσει, αλλά δεν είναι έτοιμος ο ελληνικός λαός να γονατίσει και να ταπεινωθεί. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Ο κύριος Λαμπέρς για τους πράσινους. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, τα στοιχεία για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση είναι δεδομένα χρειάζονται διαφορετικέ αλλαγέ που θα επιτρέψουν στην Ευρώπη να ξανασταθεί στα πόδια τη. Και αυτό για μένα σημαίνει μια φορολογία η οποία να είναι οικονομικά αποτελεσματική, να προστατεύει το περιβάλλον, αλλά να είναι και οικονομικά και κοινωνικά δίκαια. Πρέπει να γίνει βιώσιμο το συνταξιοδοτικό σύστημα, αλλά σεβόμενο το δικαίωμα, τα δικαιώματα των πιο ευάλωτων και πιο φτωχών. Θα πρέπει να μειωθούν οι στρατιωτικέ δαπάνε που κάνουν δυστυχώ στην Ελλάδα ένα από του πρωταθλητέ στο ΝΑΤΟ. Πρέπει να δημιουργηθεί μια αποτελεσματική δημόσια διοίκηση. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την, ε, το πελατειακό κράτος και τη διαφθορά. Το, η ελληνική κυβέρνηση ε, εξελέγει τον Ιανουάριο. Πολλές φορές αδέξια ίσως καθυστερημένα έχει μπει στο δρόμο αυτό των μεταρρυθμίσεων. Αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε επενδύσεις. Για να υπάρχει επένδυση πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις στην ελληνική οικονομία. Και ευχαριστώ τον κύριο Τίμερμανς που τόνισε ότι η Κομισιόν είναι έτοιμη να βοηθήσει. Μπορεί το Συμβούλιο να μου επιβεβαιώσει ότι η Ελλάδα είναι από τις χώρες που χρειάζονται περισσότερη βοήθεια για τις επενδύσεις. Αλλά κάτι ακόμα πρέπει να γίνει είναι να γίνει βιώσιμο το ελληνικό χρέος. Ήδη το 2010 ήταν μη βιώσιμο. Παρέμεινε μετά από το πρώτο κούρεμα και το 2012. Εξακολουθεί να είναι και τώρα μη βιώσιμο και οι διαρθωτικές αλλαγές που έχουν επιλυθεί στην Ελλάδα θα το κάνουν ακόμα λιγότερο βιώσιμο. Αυτοί οι οποίοι αρνούν να δεχτούν μία αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους δείχνουν μια τεράστια οικονομική ανικανότητα ή αλλιώς μια άρνηση της πραγματικότητας που υποκρύπτει ενοχή είτε μια ιδεολογική μονομανία να κάνει κανείς τους, ε, αυτούς που δανείστηκαν χρήματα να πληρώσουν την ύφη αφήνοντας τους δανειστές, τους άλογους δανειστές χωρίς καμία κύρωση. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν συγκεκριμένες δεσμεύσει για την αναδιάρθρωση του χρέου. Έλεγε ο Άλμπερτ Αϊνστάιν ότι ο παραλογισμό είναι να κάνει κανεί συνέχεια το ίδιο πράγμα περιμένοντα να είναι διαφορετικά τα αποτελέσματα. Ελπίζω ότι αντί για τον παραλογισμό θα επικρατήσει η συλλογική ευφυΐα στο Συμβούλιο. Ξέρω ότι σε κάποιες κυβερνήσεις δανειστών μέσα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υπάρχουν ορισμένοι που ζητούν την αποτυχία των διαπραγματεύσεων, θέλουν την έξοδο της Ελλάδος από την Ευρωζώνη. Εδώ και πολύ καιρό. Το ξέρω, έχω ακούσει να μου το λένε και προσωπικά θεωρώ ότι είναι μια ανεύθυνη στάση. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που μπορεί να ενοχλούν ορισμένους γιατί αντιτίθενται στην επικρατούσα άποψη. Αλλά δεν είναι αυτός λόγος να ανοίξουμε την πόρτα στην καταστροφή της... Ε, δεν μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε, να στιγματίζουμε τον άλλο επειδή είναι διαφορετικός και να τον καταδικάζουμε. Ευρώπη της Ελευθερίας και της Άμεσης Δημοκρατίας, ο κύριος Νούταλ. Πρόεδρε, στις ε, τελευταίες ευρωεκλογές ε, τρελαινόμασταν ε, όταν γίνονταν λόγος για Ευρωπαϊκό στρατό. Τώρα εδώ λέτε ότι ο Ευρωπαϊκός στρατός είναι ένας μακροπρόθεσμος ευρωπαϊκός στόχος πριν από το δημοψήφισμα μάλιστα μας το διευκρινίζετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πίτροπε. Πώς τώρα θα αντιμετωπίσει το θέμα της μετανάστευσης η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς θα αντιμετωπίσει το TTIP που είναι επίμαχο και φυσικά την Ελλάδα Τώρα, μετανάστευση. Ε, χτες κάποιοι Βρετανοί ε, ε, βουλευτές δεν μπόρεσαν να φτάσουν εδώ λόγω του χάους που επικράτησε στο Καλέ. Αποτέλεσμα των μεταναστών που ορμούσαν στα φορτηγά ε, προσπαθώντας να περάσουν στην Αγγλία μέχρι που έβαλαν και φωτιά. Αποτέλεσμα το τούνελ έκλεισε Υπάρχει μισό εκατομμύριο μετανάστες στη Μεσόγειο και περιμένει να έρθει στην ε, Βόρεια Ευρώπη. Και άλλο μισό εκατομμύριο περιμένει στην Αφρική. Και αυτό που είναι χειρότερο είναι ότι δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Μας λένε ότι το ISIS χρησιμοποιεί αυτό το χάος για να ε, εισάγει την διαστραμμένη του ιδεολογία στην ε, Ήπειρό μας, σε πράγμα που καθιστά την επόμενη τρομοκρατική επίθεση όχι υπόθεση του αν, αλλά του πότε και πού. Κύριε Τίμερμαντς, έχω μια καλύτερη πρόταση. Η απάντηση είναι το αυστραλιανό μοντέλο που προστατεύει τη, τα σύνορα και ένα, ένα ατσάλινο τείχος που δείχνει ότι δεν είμαστε ό,τι να είναι στην Ευρώπη. Τώρα, γιατί τι είπε και στο Στρασβούργο νωρίτερα αυτό το μήνα, ακυρώσατε την ψηφοφορία για το είπε. Εσείς ε, ε, απογοητεύσατε εκατομμύρια πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη που είχαν θεμητές προσδοκίες. Δίνει, η TTIP δίνει άδικο πλεονέκτημα στις μεγάλους ομίλους. Είναι το όνειρο κάθε λομπίστα. 30.000 λομπίστες είναι εδώ στις Βρυξέλλες, πάνω από 40 ανά ευρωβουλευτή. Περισσότεροι λομπίστες εδώ από ό,τι στη Ουάσιγκτον. Και άρα λοιπόν δεν με πλήσει που η Κομισιόν και οι μεγάλες ομάδες εδώ στο Κοινοβούλιο στηρίζουν την TTIP. Ε, ανησυχείτε για τις αρνητικές επιπτώσεις της TTIP. Θα πρέπει να βάλουμε κατά μέρο τις πολιτικές μας διαφορές, να σταθούμε ενωμένοι κατά αυτής της ε, μυστικής, ε, μυστικής, μυστικιστικής συμφωνίας. Και τέλος, πραγματικά η καρδιά μου λυπάται τους Έλληνες που γιατί βλέπω ότι το λίκνο της δημοκρατίας απειλείται από τους γραφειοκράτες και ας, ας εναντιωθούμε λοιπόν στο TTIP και σας ενωθούμε στην υποστήριξη του λαού της Ελλάδας. Σας ευχαριστώ. Για να διορθώσω κάτι, ο πρόεδρος Σούλτς είχε αποφασίσει να αναβάλει την ψηφοφορία και η σύνοδος αποφάσισε να αναβάλει τη συζήτηση. Ούτε κυρώθηκε η ψηφοφόρια, ούτε κυρώθηκε η συζήτηση. Απλώς αναβλήθησαν. Τώρα, εξ ονόματος της ομάδας Ευρώπη για την ε, ε, ε, ελευθερία, η κυρία Λεπέν. Με ψάχνετε στην πρώτη γραμμή, κύριε Πρόεδρε, σωστά, αλλά εδώ είμαι. Η δημοκρατία δύσκολα προχωράει προς τα μπρος εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατέβηκα βέβαια κάποιες θέσεις ε, θα μπορούσε να είμαι και στην πρώτη γραμμή, αλλά αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που τόσο πολύ αγαπάει τη δημοκρατία και σέβεται όλες τις ομάδες, δύσκολα θα βρει μια λύση και για μένα και να μην κάνει πια αυτό που σε όλους φαίνεται τόσο τρομερή διάκριση. Κύριε Ευρωβουλευτές, οι διαπραγματεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ελλάδα είναι σκληρές. Κανείς δεν θέλει να αφήσει τίποτα και επιβάλλεται η λιτότητα στην Ελλάδα που καταστρέφει τη χώρα. Η μείωση του ελάχιστου, σταθμού, του ελάχιστου μισθού, των συντάξεων, η αύξηση των φόρων, όλα αυτά καταστρέφουν τη χώρα και οικονομικά τους ίδιους τους πολίτες. Η Ελλάδα με 180% έλλειμμα δεν μπορεί να αποζημιώσει τους δανειστές. Αλλά ζητάτε από τους Έλληνες να εξακολουθεί να αναλαμβάνει αυτό το φορτίο, αυτού του φοβερού χρέους. Εδώ πέρα πρόκειται για σκλαβιά λόγω χρέους. Σκλαβιά για χρέος που καταργήθηκε ακόμα και πρόχριστου. Νομίζω λοιπόν ότι πάμε πάρα πολύ πίσω ότι να πηγαίνουμε μπροστά. Δεν θα μπορέσει 30 Ιουνίου να πληρώσει η Ελλάδα τους δανειστές εφόσον δεν υπάρχει συμφωνία και άρα θα πτωχεύσει. Θυμηθείτε τι ψήφισε το 2014 το Κοινοβούλιο, το ονομάσαμε το τείχος. Ήταν ένας ε, μηχανισμός. Αλλά τι θα κάνουν οι Έλληνες από τα μιευτές που τι έλεγε το κείμενο εκείνο, ότι κάτω από 100.000 ευρώ προστατεύονται από τα μιεύσεις και οι άλλες όχι. Δεν τα είπατε όμως όλα. Είπατε το άρθρο 6 του κειμένου αυτού επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μειώσει το ποσό αυτό από 100.000 σε τι, σε 20, 10.000, 5.000, 0 ευρώ. Άρθρο 6. Να σας το θυμίσω. Λέει ότι τα ποσά, οι 100.000 δηλαδή, θα αποτελέσουν αντικείμενο περιοδικής επανεξέτασης ανάλογα με την κατάσταση τροπεζικού τομέα και της οικονομικής κατάστασης της εν λόγω χώρας πριν τις 3 Ιουλίου του 2020. Ουφ, Εκτός, λέμε τα, όμως, εκτός αν υπάρξουν απρόβλεπτα γεγονότα και χρειαστεί αυτό να γίνει πιο νωρίς. Τυραννία είναι αυτή και ηλίθια μάλιστα. Όταν καταλάβουν οι Ευρωπαίοι πολίτες αυτά που κάνετε, το τραπεζικό σας σύστημα θα καταστραφεί και θα έχουμε πιο γρήγορα bank run. Το ευρώ τελικά θα οδηγήσει να καταστραφούν οι αποταμιεύσεις του κόσμου. Εσείς ψηφίσατε το κείμενο αυτό, το κρύβετε όμως στους πολίτες τι θα γίνει όταν πτωχεύσουν οι τραπεζές τους. Πρέπει να μην έχετε πια το ευρώ, να σταματήσει αυτή η τρέλα, να επανέλθουμε στη δημοκρατία και ο κάθε λαός να έχει και πάλι το εθνικό του νόμισμα. La parola all'onorevole Papadakis non iscritto. Το λίγο έχει... Να, επειδή σε βλέπα να... Είσαι αλλού.